ως τις 8 και από τις 9 έως τα μεσάνυχτα. Η ημερήσια διάταξη είναι δημοσιευμένη και στο ίντρανετ. Κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης.